μια πρόταση ψηφίσματος θα ψηφιστεί αύριο στι 12 και επίση αύριο στις 8.30 θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε μέχρι τη μία.